Συνεχίζουμε τώρα με το έργο της υποεπιτροπής μας, λέει η κυρία Βαλενθιάνου, στην Προεδρία. Έχετε την ημερήσια διάταξη. Τώρα πρέπει να περάσουμε στην γνωμοδότηση για τα αγαθά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν ε, στην εκτέλεση της θανατικής ποινής ή στο βασανισμό. Έκθεση που έχει να κάνει με την αθεώρηση του αρχικού κανονισμού του 2005. Και μετά θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο. Εγώ δεν θα μπορώ να είμαι. Θα προεδρεύσει ο κύριος Πρέντα το κομμάτι αυτό. Συνεπώς, αν δεν έχετε αλλαγέ, είμαστε στο πρώτο σημείο τη ημερήσιας διάταξη. έτσι δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε θα δώσω το λόγο στην κυρία Λόκερμπιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι η εισηγήτρια λοιπόν σε ό,τι αφορά αυτό το σύντομο γνωμοδότηση. Ε, πρόκειται για μια αρκετά τεχνική γνωμοδότηση, αλλά θα ήθελα να σας ε, τονίσω ευθύς εξ αρχής ότι αυτός ο κανονισμός κατά των βασανιστήριων είναι πάρα πολύ σημαντικός και πρόκειται για μια, ένα πολύ καινοτόμο κανονισμό τον οποίο έχουμε καθώς ε, ρυθμίζει ε, θέματα εμπορίου, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο του εμπορίου σε ανθρώπινα δικαιώματα, ειδικότερα δηλαδή σε ό,τι αφορά την εκτός της θανατικής ε, ποινής και των ε, βασανιστήριων. Νομίζω δηλαδή πως αυτό αποτελεί ε, μία απόδειξη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να υποστηριχθούν και να προωθηθούν μέσω νομοθεσίας και όχι μόνο διεθνούς συνεργασίας ε, και διαλόγου. Και όταν αυτός ο κανονισμός, ο παλαιότερος κανονισμός είχε υιοθετηθεί το 2006, είχαμε λάβει ε, αναγνώριση από τον Επιστονό των Ηνωμένων Εθνών για τα ζητήματα των βασανιστήριων. Ε, μας είπε ότι ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένο με αυτόν τον κανονισμό και κάλεσε άλλες κυβερνήσεις να αντιγράψουν ε, ένα τέτοιο νομοθέτημα στην ε, δική του εθνική νομοθεσία και ε, μάλιστα αξίωσε τη δημιουργία ενός διεθνούς νομοθετήματος. Και παρότι δυστυχώς δεν καταφέραμε να, είναι, να αναλάβει ηγετικό ρόλο, εμείς να αναλάβουμε συγγνώμη ηγετικό ρόλο και ανέλαβε τελικά η ΑΦΕΤ, θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε στο βαθμό που μπορούμε. Επίσης, Βλέπω ε, με χαρά μου πως το σχέδιο έκθεσης ε, της ε, συναδέλφου από την Αλδεμαρία ε, περιλαμβάνει πολλά στοιχεία και θετικά στοιχεία και υπάρχει και ευρεία συνένεση μεταξύ των εισηγητών για πολλά ζητήματα και ελπίζω βέβαια πως και με τους σκιώδεις εισηγητές θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια αντίστοιχη ευρεία συνένεση. Θα σας παρουσιάσω τώρα λίγο την γενική μας προσέγγιση στη συνέχεια της τροπολογίας μας. Πρόκειται λοιπόν για ένα περίπλοκο ζήτημα, όπως είπα. Πρέπει να είμαστε δηλαδή πολύ λεπτομερείς σε όλες τις τροπολογίε ε, που κάναμε ε, και στο ε, workshop το οποίο οργανώσαμε. Είχαμε μια πολύ επικοδομητική συνάντηση και εκεί η Επιτροπή, ο, ο κλάδος του εμπορίου και οι κυβερνητικέ οργανώσει είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν το ζήτημα. Επίση υπήρξε μια διαβούλευση, εκτό δηλαδή αυτού του workshop, με τις ε, δύο πηγές ε, εμπειρογνωμοσύνη, δηλαδή την Omega ε, Amnesty και την Reprieve, οι οποίε δηλαδή είναι πολύ σημαντικέ μη κυβερνητικέ οργανώσει, οι οποίε όμω υιοθετούν διαφορετικέ απόψει σε ό,τι αφορά κάποια σημαντικά ζητήματα. Και εδώ θα ήθελα να σα πω πω η Amnesty και η Omega δημοσιεύουν σήμερα τις δικές τους έδρας ε, ό,τι αφορά ακριβώς το εμπόριο τέτοιων εμπορευμάτων. Οι προτάσεις λοιπόν που γίνονται από την Επιτροπή ε, αποτελούν πραγματικά θετικά βήματα για την βελτίωση του γενικότερου πλαισίου. Ε, ήδη το σχέδιο κανονισμού περιλαμβάνει ε, ε, ε, μία σειρά από αξιώσεις από την πλευρά μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων θεσμών. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το ευέλικτο σύστημα ελέγχου, σε ό,τι αφορά ιδιωτικά προϊόντα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ε, ενέσεις ε, στο πλαίσιο θεματικών καταδικών ε, και το πώς μπορούν να προσθέτονται στην λίστα των ελεγχόμενων ειδών τέτοια προϊόντα. Εμείς λοιπόν χαιρετίζουμε τέτοιες συμπεριλήψεις και πράγματι θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα αυτά τα προϊόντα στα, στην λίστα των ελεγχόμενων προϊόντων. Ωστόσο θα θέλαμε να, ήμασταν, να είχε υπάρξει η Επιτροπή ακόμα πιο φιλόδοξη, να περιλάβει και άλλα προϊόντα και να έχει και άλλες δυνατότητες για τους πολίτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τον εμπορικό κλάδο ε, προκειμένου να μην μέσω συμμετέχουν σε ένα τέτοιο εμπόριο δηλαδή που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θανατικές ποινές ή βασανιστήρια. Αυτά σε γενικέ γραμμές και τώρα θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες από τις κύριες τροπολογίες που προτείνονται στο πλαίσιο της έκθεσης ειδικότερα σε ό,τι αφορά το στο, ε, τα, στοχευμένο end use clause, σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς ελέγχους και ε, τις, ε, τις ε, διαδικασίες υποβολής εκθέσεων ε, από την πλευρά της Επιτροπής στο πλαίσιο της τροποποίησης των παρατημάτων. Μπορούμε προφανώς ε, να αναφερθούμε σε διάφορες άλλες τροπολογίες που περιλαμβάνονται σε επικουρικές υπηρεσίες, σε τεχνική υποστήριξη, σε διαμετακομιστικό εμπόριο, σε δράσεις προώθησης, σε προϊόντων marketing και ούτω καθεξής. Ε, όμως ε, θα αναφερθώ τώρα ειδικότερα σε ό,τι αφορά αυτήν την targeted end use clause. Ε, δεν θα ήθελα λοιπόν εδώ να υποτιμήσουμε τη δημιουργικότητα εντό εισαγωγικών ορισμένων εμπορευομένων, ειδικότερα όταν υπάρχει η ε, ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση για τέτοιου είδους προϊόντα από αντίστοιχους φορείς. Όταν δηλαδή υπάρχει, μπορεί να υπάρξει μια ε, πρόβλεψη εκ των προτέρων ή ε, ένας μηχανισμός ε, άμεσης αντίδρασης θα είναι ακόμα καλύτερο, ούτως ώστε να περιλαμβάνονται γρήγορα στη λίστα τέτοια προϊόντα. Και η πρόταση της Επιτροπής για συμπερίληψη ενός τέτοιου μηχανισμού είναι πολύ θετική. Ωστόσο γνωρίζουμε, με βάση τη δική μας εμπειρία, ότι η επιτροπή ε, και η ευελιξία είναι δύο έννοιες λίγο θα λέγαμε ασύμβατες. Άρα λοιπόν θα ε, πρέπει να ε, υπάρχει μια διαδικασία επίγουσα η οποία θα διέπει τέτοιου είδους προϊόντα και βέβαια μια τέτοια προσέγγιση δεν είναι καινοτόμα. Το Κοινοβούλιο και κατά την, το σχέδιο έκθεσης για τα βασανιστήρια έχει ζητήσει να συμπεριληφθεί μια τέτοια ρήτρα ε, μια τέτοια ρήτα υπάρχει ε, για παράδειγμα και στο πλαίσιο της ομάδας ε, της Αυστραλίας όπου περιλαμβάνονται όλα τα μέλη μας που ασχολείται με τα ζητήματα πυρηνικά και βιολογικές, πυρηνικές και βιολογικές ουσίες και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν υποστηρίξει την εισαγωγή μιας τέτοιας ρήτρας εδώ και πολλά χρόνια και η συγκήτρια υποστηρίζει λοιπόν την θέσπιση μια τέτοια ρήτρας. Εκείνη αναφέρεται σε αυτή τη ρήτρα ως catch all clause, εμείς αναφερόμαστε σε αυτήν ως ε, targeted end use clause. Ε, μας δίνει τη δυνατότητα, στα κράτη-μέλη δηλαδή, να ε, εφαρμόζουν μια γενικότερη ε, Ε, και τους επιτρέπει στοχευμένα ε, να ε, προβαίνουν ε, για παράδειγμα στην διακοπή μια τέτοια ε, διαμετακόμιση ενό εμπορίου, όχι όταν περιλαμβάνεται το συγκεκριμένο εξάρτημα στην λίστα των ελεγχόμενων προϊόντων, αλλά όταν υπάρχει μια υποψία ότι αυτή, αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο. Επίση, στην ίδια ρήτρα αναφέρεται ότι θα πρέπει να αναφέρονται σαφεί λόγοι από την πλευρά των κρατών μελών. Και αυτό το κάνουμε για να διασκεδάσουμε τι ανησυχίε ότι θα μπορούσαν τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν αυτή τη ρήτρα κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Ε, υπάρχει δηλαδή ε, ανάγκη συντονισμού μεταξύ Επιτροπή και κρατών μελών, ώστε ακριβώ να γίνεται ορθή χρήση τη εν λόγω διάταξη. Επίση, ε, προτείνουμε η Επιτροπή να αποφασίζει κατά πόσο τα εν λόγω αγαθά θα πρέπει να προστίθενται μετά στο σχετικό παράτημα ή όχι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους εθνικούς ε, πολιτικούς μηχανισμούς. Ε, η πρόταση της Επιτροπής για ενίσχυση ε, των ελεγχών στο διαμετωπιστικό εμπόριο, ειδικότερα των ιατρικών προϊόντων, είναι πολύ θετική, αλλά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητα των κρατών να προβαίνουν σε αποτελεσματικούς ελέγχους και να αντιλαμβάνονται τις συμβατικές συμφωνίες των φαρμακευτικών εταιριών. Άρα λοιπόν εμείς προτείνουμε να υπάρχει δυνατότητα ενός εξωτερικού ελέγχου ώστε να προσδώσουμε μία ακόμα, ένα ακόμα επίπεδο ελέγχου. Άρα λοιπόν η εν λόγω τροπολογία, τροπολογία 12, ε, προσπαθεί να δώσει ε, τη δυνατότητα στα, ε, στους, στα όργανα με τη μεγαλύτερη εμπειρογνωμοσύνη των κρατών μελών να έχουν πρόσβαση ακριβώς σε αυτές τις ε, συμβάσεις ε, των φαρμακευτικών ε, εταιριών για παράδειγμα θα μπορούσαν αυτοί οι αρμόδιοι φορείς να είναι εκείνοι που είναι αρμόδιοι για τους σχετικούς μηχανισμούς καταπολέμησης των βασανιστήριων. Ήδη δηλαδή τέτοιου είδους μηχανισμοί υπάρχουν στα κράτη-μέλη και θέλουμε η πρόσβαση σε λόγο πληροφορίες να είναι δυνατή και για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ανάλογα δηλαδή με το που αυτές δρέμουν φυσικά και θα ήθελα να τονίσω πως οι δύο ε, μη κυβερνητικέ ε, ε, οργανώσεις δεν είναι με τη στενή, του, έννοια του όρου μη κυβερνητικέ, καθώς υπάγονται ήδη σε εθνικούς ελέγχους και είναι αρμόδιες για την εξέταση των παραβιώσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες της. Αποτελούνται συνήθως από εμπειρογνώμονες οι οποίοι έχουν ακριβώς την την απαιτούμενη τεχνογνωσία και θεωρώ ε, πως θα ήταν ε, μια ε, πολύ θετική συμβολή από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η υποστήριξη αυτή τη τροπολογία. Επίση, ό,τι αφορά τώρα την υποβολή εκθέσεων, εμεί θέλουμε να μα προβλεπ... υποβάλει ετησίω η Επιτροπή στα Μελ μία ετήσια έκθεση σύνθεση. Μέχρι στιγμή αυτό το... η υποβολή των εκθέσεων είναι πολύ δύσκολη. Δηλαδή, η πρόσβαση στις εκθέσεις είναι δύσκολη και υπάρχει και μια ε, ε, δυσκολία σε ό,τι αφορά το συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών. Ε, η υποβολή όμως τέτοια ετήσια έκθεση ε, θα υποστήριζε και την διαφάνεια και την υπευθυνότητα και θα έδινε περισσότερες, θα ενίσχυε περισσότερο τον ελεκτικό ρόλο τη Επιτροπή. Από εκεί και μετά υπάρχουν κάποιες τροπολογίες σε ό,τι αφορά τα, το παράτημα 2 και το παράτημα 3. Εκεί λοιπόν έχω συμπεριλάβει εδώ μία σειρά από ε, ε, αγαθά ε, στις λίστες ελέγχου και στις λίστες απαγόρευσης. Και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις έχουν αναφέρει πολύ καλούς λόγους για κάθε ένα από αυτά τα αγαθά. Γιατί δηλαδή θα πρέπει να απαγορευτούν να αναφέρουν συγκεκριμένα παραδείγματα όπου έχουν χρησιμοποιηθεί και για λόγους εκτέλεση θανατικών ποινών και βασανιστήριων ή αποκλειστικά για αυτούς τους λόγους. Τώρα, έχω εδώ ε, μπροστά μου τα λεπτομερή στοιχεία, στοιχεία και για όλες τις υπόλοιπες τροπολογίες, αλλά νομίζω πως θα ήταν καλύτερο να σταματήσω εδώ ε, και να επιτρέψω στους σχεδόν συζητητές να, να θέσουν τα ερωτήματά τους. Προφανώ η συνάντηση που θα έχουμε με του κοιόδη συζητητέ ε, θα προβούμε σε μια πιο ει βάθο συζήτηση όλων των τροπολογιών και ε, παρότι θα μπορούσα να έχω συμπεριλάβει εδώ ε, να έχω υποβάλει δηλαδή περισσότερες ε, τροπολογίες, βρίσκομαι ακόμα εν αναμονή ε, κάποιων εκθέσεων από εμπειρογνώμονες. Δεν μπορώ λοιπόν ακόμα να συζητήσω τέτοιου είδου τροπολογίε. Για παράδειγμα, ε, ένα από αυτά τα ζητήματα είναι η δυνατότητα ελέγχου σε ό,τι αφορά ιατρικά προϊόντα, όπω επίση και το ζήτημα τη τροποποίηση τη λίστα των χωρών ε, στο παράδειγμα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λόχμπιλερ. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε λίγο χρόνο για συζήτηση σήμερα, αλλά οι συναντήσει των σκιωδών με την κυρία Λόχμπιλερ μπορεί να βοηθήσει για περισσότερε ε, συζητήσει σε βάθο οι σκιώδεις, έτσι. Τώρα, ο κύριος Τζιλ που είναι ένας από τους σκιώδεις. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, θέλω να σας πω ότι η... τα σχόλια των σκιωδών εισηγητών ε, δεν μπορώ να τα παρουσιάσω όλα. Εγώ αντικαθιστώ την σκιώδη τη ομάδα μου. Πρώτα απ' όλα, εκ μέρου λοιπόν τη συναδέρφου, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Λόχ Μπίλερ για την ε, έκθεση που προετοίμασε για ένα θέμα δύσκολο, ένα θέμα το οποίο επανέρχεται και επανέρχεται στις εργασίες της Υποπιτροπής μας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι πολύ ιδιαίτερο θέμα γιατί πρόκειται για αγαθά τα οποία έχουν ε, διπλή χρήση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καλό και για κακό σκοπό. Πάντα υπάρχει τεχνική πρόοδος, αυτή δεν σταματάει ποτέ. Οπότε εκ μέρου τη συναδέρφου και όδου θέλω να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο ως υπεύθυνο παράγοντας για την καταπολέμηση της θανατικής ε, ποινή και των βασανιστήριων της πρακτικής αυτής. Οι δράσεις μας λοιπόν πρέπει να συνεχιστούν και ό,τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να ενημερώσουμε τον ε, σημερινό κανονισμό πρέπει να γίνει. Το διεθνές εμπόριο επίσης αλλάζει. Υπάρχουν νέα προϊόντα, φαρμακευτικά κυρίως, και γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε σαφείς κανόνες που να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις προκλήσεις του σημερινού κόσμου. Πρέπει επίσης να προωθήσουμε τις ανταλλαγές πληροφοριών. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, μας βοηθάει να εφαρμόζουμε τον κανονισμό πιο αποτελεσματικά. Όσον αφορά τις τροπολογίες, αυτές αυτό ακριβώς κάνουν, αυτό ακριβώς αναφέρουν, ότι έτσι μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Θέλω επίσης να διευκρινίσω και τον ορισμό του όρου βασανιστήριο. Για τις άδειε εξαγωγής χρειαζόμαστε ένα πιο σαφή ορισμό, ώστε οι κανόνες που εφαρμόζονται στις εξαγωγές εφαρμόζονται πιο αποτελεσματικά. Επίσης, τα προϊόντα τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα 3 πρέπει πάντα να επιτρέπεται να εξάγονται, αλλά η άδεια αυτή δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται εφόσον τα προϊόντα αυτά βρίσκονται μέσα στον τελωνιακό χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο όταν φεύγουν από τον χώρο αυτό απαιτείται η άδεια. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις της Κιόδους εισηγήτριας για την γνωμοδότηση αυτή που ετοίμασε η συνάδελφος Λοχμπίλερ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ροντρί... Euh, Θα μιλήσω πορτογαλικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έγγραφο που μας ε, υπέβαλε. Είχαμε ε, δύο τροπολογίες σε σχέση με την επίβλεψη, την ομάδα επίβλεψης για την εφαρμογή αυτής της έκθεσης. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο είναι πολύ δύσκολο να έχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες και εγώ είχα μεγάλη δυσκολία, συγχαρητήρια όμως, είναι εξαιρετικό το έγγραφο. Μόνο κάτι υπάρχει το οποίο δεν κατάλαβα καλά και θα ήθελα περισσότερες διασαφήσεις στο 16 που μιλάμε για την εφαρμογή και την εποπτεία του κανονισμού. Ίσως τα τρία χρόνια είναι πολύ μεγάλο χρονικό περιθώριο για την εφαρμογή του κανονισμού. Ίσως θα έπρεπε να δούμε κατά πόσο δεν θα ήταν δυνατόν να ε, περιορίσουμε το χρονικό διάστημα σε δύο χρόνια και όχι τρία για να έχουμε πρόσβαση Ο συνάδελφος μίλησε για τα άρθρα που ενδεχομένως δεν θα χρησιμοποιηθούν. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορεί να γίνει θετική χρήση και με βάση τις τεχνολογίες έχουμε κάτι το οποίο όμως δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Θα ήθελα να συγχαρώ και πάλι την εισηγήτρια γιατί πρόκειται για μια δύσκολη εργασία σχετίζεται με πολλά πράγματα σε επίπεδο εμπορίου, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει σαφή θέση, δηλαδή θα πρέπει να ξέρουμε κατά πόσο ε, αυτά τα αγαθά, αυτά τα εμπορεύματα ε, μεταφέρονται και θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις προς τις χώρες που χρησιμοποιούν αυτά τα εμπορεύματα, αυτά τα είδη για βασανιστήρια και για τη θανατική ποινή. Ευχαριστούμε. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Πράγματι, είναι ένα πολύ σημαντικό και τεχνικό θέμα και δύσκολο. Γι' αυτό και θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Μπάρμπαρα, την εισηγήτρια. Πολύ σημαντική η δουλειά που έκανες. Ξέρω πόσο σοβαρά το έχεις πάρει, ξέρω ότι και τεχνικά έχεις ενημερωθεί. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Νομίζω ότι έχουμε τον ίδιο στόχο. Η τροπολογία 9 όμως με κάνει να θέλω να ρωτήσω κάτι. Γιατί καταλήγει σε μία πρόταση για ρήτρα για χώρες για μια μονομερή αντιμετώπιση, δηλαδή να μπορούν μονομερώς κάποιες χώρες να μπλοκάρουν ένα προϊόν. Αλλά αυτό πρέπει να γίνεται εφόσον ε, ξέρουμε ότι απευθύνεται σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη θανατική ποινή ή με τα βασανιστήρια. Αυτό είναι κάτι που μου θυμίζει το λεγόμενο Targeted End Use Mechanism Πρόκειται για ένα έγγραφο και η Διεθνής Αμνηστία έχει μιλήσει γι' αυτό. Κάτι το οποίο μπορεί κανείς να βρει σήμερα εύκολα. Όσον αφορά τα φάρμακα τώρα, ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα γιατί μπορεί έτσι να παγορευτούν κάποια, κάποιες ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στην αναισθησία. Γι' αυτό λοιπόν στις 23 Απριλίου είχαμε την ακρόασή μας και ακούσαμε και τους εμπειρογνώμονες οι οποίοι είναι υπέρ ενός αποτελεσματικού ελέγχου εξαγωγών βέβαια ώστε τα φάρμακα τα οποία χρειάζονται να μπορούν να κυκλοφορήσουν, να διασφαλιστεί η κυκλοφορία αυτή. Από την άλλη μεριά όμως τα ευρωπαϊκά φάρμακα να μην φτάνουν στις αίθουσες όπου εκτελούνται οι θανατικές ποινές. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί. Και εντάξει, μπορεί να μην είναι τέλεια, αλλά νομίζω ότι είναι μια αναλογική απάντηση που δίνουμε, ανάλογα με το πρόβλημα δηλαδή η απάντηση που δίνουμε με την πρότασή μας αυτή. Θέλω λοιπόν να μάθω από την Μπάρμπαρα, είναι διατεθειμένη να αποκλείσει τα φάρμακα αυτά από την ρήτρα ασφάλειας. Δεύτερη παρατήρηση. Οι τροπολογίες 2, 3, 5, 9, 10, 15 και 16 του σχεδίου γνωμοδότησης είναι ίδιες, νομίζω εγώ. Ή επικαλύπτονται με τροπολογίες της συναδέλφους Χάκε στην Επιτροπή Ίντα, που είναι η επί της συναδελφου χακε στην επιτροπη ιντα που ειναι η επι της αρμοδια Συμφωνεί, συμφωνείς Βάρβαρα. Μπορεί να αποσύρεις κάποιες τροπολογίες, πώς το βλέπεις εσύ. Δεν έχω χρόνο για να δώσω σε άλλο το λόγο πέρα από την εισηγήτρια. Η εισηγήτρια μόνο γιατί αρχίζουμε να τρώμε από το χρόνο που είχε προβλεφθεί για την επόμενη συζήτηση. Οπότε παρακαλώ κυρία Λόχμπίλερ να απαντήσετε όσο γίνεται πιο γρήγορα και ζητώ συγγνώμη στους υπόλοιπους που ήθελαν να πάρουν το λόγο. Δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς και οι σκιώδες εισηγητές με την εισηγήτρια μπορούν να συνεχίσουν να δουλεύουν τις επόμενες ημέρες. Μπάρμπαρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για όλα τα σχόλια που ακούσαμε. Θα απαντήσω μόνο στα ερωτήματα που τέθηκαν. Κυρία Ροντρίγκε, στην τροπολογία 16 ε, Αναφέρθηκα λοιπόν εδώ σε τρία έτη με βάση το πλαίσιο διπλής χρήσης, το Dual Use Framework, αλλά θεωρώ πως αυτό ε, οφείλεται σε περιπλοκές κατά την υποβολή των εκθέσεων, αλλά μπορούμε να το ξανακοιτάξουμε. Τώρα, ε, από την πλευρά ε, του ε, ε, τα σχόλια. Νομίζω πως εδώ χρειαζόμαστε ε, πιο εκτενή συζητήσεις, οπότε μπορούμε να το κάνουμε στο πλαίσιο της συνάντησης των σκιωδών εισηγητών. Τώρα, Μαρκ, αναφέρθηκε σε ένα ζήτημα σε ό,τι αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση θανατικών, καταδικών, θανατικών ποινών. Ε, αυτό από μόνο του ο ζήτημα αποτελεί ε, ε, πρόβλημα, γιατί οι εμπειρογνώμονες από την κοινωνία των πολιτών έχουν δύο διαφορετικές απόψεις ως προς το ποια είναι η βελτιστή πρακτική. Εγώ αυτό που λέω είναι να αναβερόμαστε σε ε, προϊόντα που σχετίζονται με την ασφάλεια στο πλαίσιο αυτής της διάταξης, όχι σε φαρμακευτικά προϊόντα. Και αυτό ε, γιατί ένα από τα επιχειρήματα το οποίο θεώρησα πιστικά από, αυτό, από αυτούς που υποστηρίζουν να μην ε, υπευθύνουν. Ε, ε, για παράδειγμα η γερμανική εταιρεία η οποία, η οποία παράγει τέτοιου είδους φαρμακευτικά συσκευάσματα, μια γερμανική που για παράδειγμα, τις οποίες τα προϊόντα χρησιμοποιούνται για την, ε, ε, ε, ε και στο Μιζούρι, χρησιμοποιούνται και για αναισθητοποίηση. Οπότε, αυτό που έχει, έχει ε, γίνει είναι όταν γίνεται μια πώληση αυτών των φαρμάκων στις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε τα εν λόγω φαρμακεία, ας δεν μπορούν να, να πουλήσουν αυτό το φάρμακο, για παράδειγμα, σε φυλακές. Για υπήρξε μια τέτοια περίπτωση όπου δηλαδή ε, προσπάθησε ε, μια, δηλαδή να κάνει μια τέτοια αγορά και ε, δεν ήταν δυνατό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα, κατά την, μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτό και κατά την συνάντηση των αστιωτών εισηγητών. Ε, πρόεδρε, μπορώ να ρωτήσω πότε θα είναι η πρώτη συνάντηση αυτή. Όχι, δεν έχουν ορίσει καν οι πολιτικές ομάδες ακόμα τους σκιώδεις τους. Η Γκουε, για παράδειγμα, δεν έχει ορίσει σκιώδη. Είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε αυτό. Ελπίζω τις επόμενες ημέρες η γραμματεία θα φροντίσει να επιμείνει ώστε να μας έρθουν τα ονόματα των ε, σκιωδών που λείπουν. Ήρθε κάποιος από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και εφόσον ήρθε θα του δώσω το λόγο και ειλικρινά λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπορούμε να χειριστούμε το χρόνο με μαγικό τρόπο για να έχουμε περισσότερο. Έχουμε αυτό που έχουμε. Οι διατάξεις δεν λαμβάνουν πάντα υπόψη το χρόνο. Έτσι κι αλλιώς είχαμε τον πρόεδρο της Τινησίας που άργησε. Έχουμε και τη συζήτηση για την Αίγυπτο μετά. Μια που ήρθατε, πάντως σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Θα σας δώσω το λόγο και για άλλη μια φορά ζητώ συγνώμη στους προσκεκλημένους μας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Με την άδειά σας, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλω να πάρω το λόγο είμαστε αρμόδιοι για την εξωτερική πολιτική όσον αφορά το θέμα αυτό. Δεδομένου λοιπόν του γεγονότος ότι έχουμε πολύ λίγο χρόνο, θα απαντήσω πάρα πολύ σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Λόκβιλερ πρώτα απ' όλα, την εισηγήτρια, για τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασε το σχέδιο γνωμοδότησης. Θέλω επίσης να πω ότι υπάρχουν διάφορες τροπολογίες με τις οποίες μπορεί να συμφωνήσει εν μέρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 3, 4, 15 και 16. Και συμφωνούμε κυρίως με τη 15 που αναφέρεται στο συντονισμό, μια ομάδα συντονισμού για την ε, ρύθμιση, όπως είχαμε για την ε, καλή χρήση των ελέγχων εξαγωγών πιστεύουμε ότι η κατεξοδότηση αρμοδιότητες που έχουν δοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια τέτοια ομάδα συντονισμού θα μας οδηγήσει σε καλύτερη εφαρμογή του κανονισμού. Ένα πράγμα έχω να προσθέσω για την τροπολογία που προτείνεται όσον αφορά τη λεγόμενη Targeted End Clause, που δεν στηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό συμβαίνει για τους εξής λόγους. Εμείς πιστεύουμε ότι η τροπολογία βάζει εδώ πέρα διάφορα νομικά ζητήματα. Πιστεύουμε ότι η εισαγωγή ε, μιας τέτοιας ε, ρήτρας ε, τελικής χρήσης δεν συνάδει με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε με την ε, Γενική Συμφωνία Δασμών. Ο κανονισμός αναφέρεται σε αγαθά τα οποία δεν έχουν στρατιωτική χρήση. Γι' αυτό υπάρχει και διάκριση με τον κανονισμό για τα βασανιστήρια. Τέτοια ε, αγαθά χρησιμοποιούνται σύμφωνα με αυτή τη διάταξη και για στρατιωτικούς και για μη στρατιωτικούς λόγους. Οποιαδήποτε στρατιωτική χρήση δεν δικαιολογείται βάσει του 21.5 της Συμφωνίας ΓΚΑΤ και έτσι ισχύουν οι περιορισμοί των χωρών μελών που έχουν να κάνουν με το 346 1β της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν η ρύθμιση για χρήση βασανισμών πρέπει να δικαιολογείται από το άρθρο 21b. Πρέπει να προστατεύεται η ηθική και η ανθρώπινη ζωή και υγεία. Πρέπει να χρησιμοποιούνται με τρόπο που να μην γίνεται διάκριση σε βάρος χωρών όπου ισχύουν κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι λαμβάνοντας υπόψη τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συμφωνία ΓΚΑΤ, ο 1236 του 2015 πρέπει να θέτει ομοιόμορφους κανόνες και όλες οι ρήτρες τελικής χρήσης λοιπά να επιτρέπουν στις χώρες μονομερώς να αποφασίζουν για, το, για την τελική χρήση των προϊόντων. Όπως προτείνεται στην τροπολογία 15, είναι κάτι που δεν μπορούμε να δεχτούμε. Οι ομοιόμορφοι κανόνες πρέπει να έχουν την εξή μορφή. Είτε εκ των προτέρων άδεια για όλα τα προϊόντα, η μη εκ των προτέρων άδεια πάλι για όλες τις εξαγωγές όλων των προϊόντων. Δεν υπάρχει ειδική διάταξη όσον αφορά την εμπορική πολιτική που να λέει ότι ελεύθερα εξάγονται σε άλλες χώρες και το τρίτο είναι ότι για οποιονδήποτε εξαγωγέα ή transit ο φορέας ο ενδιάμεσος είναι υπεύθυνος για το κατά πόσο υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα αυτά για θανατική ποινή, βασανιστήρια κτλ. Αυτές ήταν κάποιες σκέψεις που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας για την τόσο σημαντική ε, τροπολογία που προτείνετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λοκβίλερ. Θέλετε κάτι να πείτε. Δεν έχω να πω ε, πολλά. Ε, ε, και ε, λυπάμαι ε, για το γεγονός ότι το, η γραμματεία δεν κατάφερε να μου διασφαλίσει να υπάρξει μια γνωμοδότηση και από την νομική υπηρεσία του Συμβουλίου. Ευχαριστούμε κυρία Λόχ Μπίλερ. Φαντάζομαι θα την έχετε την νομική γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προφανώς και την χρειάζεστε για να συντάξετε τη γνωμοδότησή σας. Χρειαζόμαστε την νομική γνωμοδότηση από την νομική υπηρεσία. Καλώς, σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω 2 Ιουνίου, που είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών, να φτάνει. Τώρα, αν κάποιος από την ΚΟΕ είναι σκιώδης, να μας το πείτε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πρεντά τώρα θα προεδρεύσει και περνάμε στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αίγυπτο. Ε, ε, Καλημέρα σε όλους σας. Θα αρχίσουμε τη συζήτηση αυτή, την ανταλλαγή αυτή απόψεων όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο. Πρέπει εδώ να διαπιστώσω ότι από τους 31 που είναι κανονικά τα μέλη της Επιτροπής μας, έχουμε μόνο τέσσερις παρόντες. Εγώ και άλλοι τρεις. Είναι θλιβερό. Κυρίως γιατί έχουμε συζητήσει πάρα πολύ προετοιμάζοντας αυτή την ανταλλαγή απόψε. Όταν το συζητάγαμε και το προετοιμάζαμε, ήταν πολύ περισσότεροι οι παρόντες. Και είδαμε και πάθαμε να οργανώσουμε την ανταλλαγή αυτή. Τέλος πάντων, το. Το καταγγέλω αυτό, τι να πω. Αρχικά θα ερχόταν εδώ ο κύριος Καγιέκ, που είναι ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Αιγύπτου. Κανονικά θα ερχόταν να συμμετάσχει στην ανταλλαγή αυτή απόψεων, αλλά με θλίψη μάθαμε ότι δεν μπόρεσε τελικά να έρθει. Η, η υποεπιτροπή μας υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα με μια ισχυρή εντολή που μας επιτρέπει να έχουμε τις επαφές αυτές. Κρίμα λοιπόν που ο κύριος Σφαγέκ δεν μπόρεσε να ταξιδέψει και να έρθει. Μια τέτοια ανταλλαγή απόψεων την είχαμε με υπεύθυνους από αντίστοιχα όργανα. Τώρα, για την Αίγυπτο πιο συγκεκριμένα, φυσικά τις, τον τελευταίο καιρό συζητάμε πάρα πολύ για το θέμα της ασφάλειας, για τον ρόλο της Αιγύπτου επίσης στην αντιπαράθεση που υπάρχει με τους ριζοσπάστες οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο την ίδια την ασφάλεια. Από την άλλη μεριά βέβαια, και αυτό ακριβώς είναι το διακύδευμα της σημερινής μας συνάντησης και συζήτησης, θέλουμε να συζητήσουμε για τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα, την ειρηνική λύση, την κοινωνία των πολιτών, την ελευθερία των δημοσιογράφων και πιο συγκεκριμένα για στρατιωτικές δίκες που γίνονται και όπου δικάζονται εκεί μη στρατιωτικοί. Για παράδειγμα, έξι νέοι ε, εκτελέστηκαν και πάνω από 100 έχουν καταδικαστεί, μεταξύ άλλων ο πρόεδρος Μόρση. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να υπενθυμίσουμε στις αρχές της Αιγύπτου την έκκληση που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ξανά και ξανά προκειμένου να μην εκτελεί τη θανατική ποινή, που είναι μια πάγια θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζουμε ξανά και ξανά την ε, θέση μας αυτή. Είμαστε κατά της θανατικής ποινή έτσι κι αλλιώς και όπου προβλέπεται από την νομοθεσία ζητάμε από όλες τις χώρες αυτές να δεχτούν μια συμφωνία προκειμένου να μην εκτελεί τη θανατική ποινή. Και όσον αφορά τις καταδίκες, τις μαζικές, έχουμε πει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε διάφορα ψηφίσματά μας το έχουμε συμπεριλάβει, ότι οι μαζικές αυτές καταδίκες έρχονται σε αντίθεση με τις διεθνείς υποχρεώσεις χωρών όπως η Αίγυπτος και είναι και σε αντίθεση με το ίδιο το πνεύμα του κράτους δικαίου. Αυτά είναι τα θέματα που απασχολούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα λοιπόν, πάντα για την Αίγυπτο πρέπει να αναφερθούμε και στο ζήτημα της κατάστασης των γυναικών και των κοριτσιών στην Αίγυπτο. Υπάρχει η απειλή για σωματική και σεξουαλική βία σε βάρος τους και στο δημόσιο χώρο και ιδιωτικός. Ελπίζουμε η Αιγυπτιακή κυβέρνηση να καταργήσει τους νόμους αυτούς που στηρίζει τέτοιες πρακτικές φυσικής και σεξουαλικής βίας σε βάρος των γυναικών προκειμένου να συνάδει με το διεθνές δίκαιο και με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά όσον αφορά λοιπόν τις γυναίκες και τα κορίτσια στην Αίγυπτο. Αυτά εισαγωγικά. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους τον κύριο Χαφές Ζαμπού Σεντά, ο οποίος είναι πρόεδρος της Αιγυπτιακής Οργάνωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και επίσης τον κύριο Μπαχέι Ελντίν Χασάν, που είναι διευθυντής και ιδρυτής του Ινστιτούτου του Καΐρου για μελέτες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και οι δύο, μάλλον ο καθένας τους, έχει 10 λεπτά στη διάθεσή του, προκειμένου να μας παρουσιάσετε την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο, έτσι όπως εσείς τη βλέπετε. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι που ήρθατε και έχετε το λόγο. Πρώτο κύριο Χαφέ Σαμπού Σέντα, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ε, θα ήθελα να στήσω ε, συγγνώμη που δεν ήταν εδώ ο συνάδελφος επειδή είχε κάποια άλλη υποχρέωση. Είναι πραγματικά θετικό το ότι με βρίσκομαι εδώ γιατί εκπρόσωπο με ομάδα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά συμμετέχω και στο Εθνικό Σύμβουλο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Και θα ήθελα να σας ε, διαβεβαιώσω ότι όλοι ε, έχουμε τις ίδιες ε, αρχές σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλοι μας αγωνιζόμαστε για, την, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αίγυπτο ε, δηλαδή και στις 25 και στις 3 Ιουνίου ε, οι επαναστάτησεις ε, οδήγησαν σε νέες ελπίδες σε ό,τι αφορά την δημιουργία μιας δημοκρατίας και ενός κράτους δικαίου που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελπίζουμε πως θα καταφέρει ο λαός μας να επιτύχει αυτούς τους στόχους. Κατά την παρέμβασή μου θα αναφερθώ σε τρία ζητήματα. Καταρχήν θα αναφερθώ στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ε, κοινωνία στην Αίγυπτο. Ε, μετά από τις 3 Ιουνίου όλοι γνωρίζετε ότι βρισκόμαστε σε μια τέτοια μεταβατική ε, περίοδο. Και η επιμέρους πρόκληση είναι ο τουρισμός. Μετά, δεύτερο θα αναφερθώ στο μέλλον της Αιγύπτου και ειδικότερα δύο τεινά εδώ. Πρώτον το νέο σύνταγμα και από εκεί και μετά οι συστάσεις ε, που έγινε από το Εθνικό Συμβούλιο στη Γενέβη προς την κυβέρνη μας ε, και ε, το τρίτο ζήτημα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι η θανατική ποινή και νομίζω εδώ πως όλοι μας ως υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουμε την κατάργηση της θανατικής ποινής και οι ακτιβιστές στην Αίγυπτο εργάζονται επί αυτού του ζητήματος εδώ και πολύ καιρό και ε, πριν από μία εβδομάδα υπήρξε μία πρόταση από το Εθνικό Συμβούλιο ε, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, για να ζητηθεί από την κυβέρνηση να απαγορευτεί η επιβολή της θανατικής ποινής γιατί ακόμα δεν έχουμε μια οριστική θανατική ε, καταδίκη του κύριου Μόση και των υπολείπων ε, της αδελφότητας, δηλαδή πρέπει να περάσει ακόμα από το μεγάλο μόφτη, οπότε ελπίζουμε πως εκεί δεν επιβληθεί σε αυτό το επίπεδο πλέον η θανατική ποινή, αλλά πρόκειται βέβαια και για μια πιο ε, μια, μια διαδικασία που είναι ιδιαίτερα μακροβία. Τώρα, να αφαιρθώ στο πρώτο από τα ζητήματα. Ε, καταρχήν τη μήνυ πρόκληση σε ό,τι αφορά το τον, ε, την ε, τρομοκρατία. Μετά από τη σύλληψη λοιπόν ε, του κυρίου Μόρση και την, το τέλος της ε, αδελφότητας υπήρξε ένα μεγάλο κύμα τρομοκρατίας παρότι δηλαδή της ε, του Αιγυπτιακού λαού για δημοκρατία μετά από, την, από το τέλος της κυριαρχίας του κυρίου Μουμπάρακ ε, ο κύριος Μόρση αναλαμβάνοντας δηλαδή τα ενία της χώρας υιοθέτησε μια πάρα πολύ αντιδημοκρατική ε, στάση. Η ε, μουσουλμανική αδερφότητα δηλαδή και ο κύριος Μόρση προσπάθησαν να επιβάλλουν μια, ένα θεοκρατικό ε, σύστημα καθεστώς ε, στην Αίγυπτο το οποίο περιθωριοποιεί όλες τις ε, θρησκευτικές μειονότητες και προσπαθεί να έχει το μονοπόλιο σε πολιτικό επίπεδο της πολιτικής θρησκείας. Και όταν υπήρξε βέβαια ε, υπήρξε αντίδραση από την πλευρά ε, του Αιγυπτιακού λαού χρησιμοποιήθηκαν εναντίον τους ε, και ρητές απειλές αλλά και θανάσιμη βία ειδικότερα μετά από, μια, από ένα συνταγματικό ψήφισμα το οποίο έδωσε απόλυτη εξουσία στον κύριο Μόρση στα τέλη του 2012. Και βέβαια για μία ακόμα φορά στις 3 Ιουνίου κατέβηκε ο λαός ε, στον δρόμο για να ε, διορθώσει, να προσπαθήσει μία ακόμα φορά να διορθώσει την κατεύθυνση που ακολουθούσε ε, η χώρα μετά από, και από την πρώτη επανάσταση. Άρα λοιπόν κατέβηκαν για μία ακόμα φορά οι Αιγύπτιοι ε, ε, Αιγύπτιοι πολίτες ε, στο δρόμο στι 3 Ιουνίου του 2013 αξιώνοντα την παρέτηση του κυρίου Μόρση όπως είχαν κάνει προηγουμένω και με τον πρόεδρο Μουμπάρακ. Ο Μουμπάρακ τότε είχε παρετηθεί αλλά ο κύριος Μόρση αρνήθηκε να το κάνει. Και ο κύριος Μόρση ήταν ξεροκέφαλος, ας το πούμε έτσι, όπως ήταν και ο κύριος ε, Ομπάραχ, ε, αρνήθηκε να παραιτηθεί και έτσι οδηγηθήκαμε σε διάφορες ε, βίες συγκρούσεις, σε διάφορα μέρη της χώρας, τα οποία οδήγησαν στο θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Σε, αντιδρώντας λοιπόν στις αξιώσεις του λαού για την καθαίρεση του κυρίου Μόρση το, οι ένοπλες δυνάμεις παρενέβησαν σώνοντας την χώρα μάλιστα από ένα ενδεχόμενο ε, εμφύλιο πόλεμο. Ε, και στις 20 ε, Ιανουαρίου είχε συμβεί ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ε, όταν κατέβηκε ο δρόμος, είχαν κατέβει τα πλήθη τους δρόμους και για δεύτερη φορά στις 3 Ιουνίου και πάλι οι ένοπλες δυνάμεις πήραν το μέρος του λαού. Μετά λοιπόν από την καθαίρεση του κυρίου Μόρση και της μουσουμανικής ε, αδελφότητας ε, ξεκίνησαν από την πλευρά τους ε, μία σειρά από τρομοκρατικές δράσεις που οδήγησαν στον, στην θάνατο εκατοντάδων προσωπικών ασφαλείας, μελών των ενόπλων δυνάμεων. Είχαμε για παράδειγμα βομβιστικές επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια, δολοφονίες αστυνομικών, εμπρισμούς και άλλου είδους ε, ζημιές ε, κτίρια αποδομής τα οποία όλα έχουν ε, τεκμηριωθεί από την, έχουν τεκμηριωθεί όντως από την Αιγυπτιακή Οργάνωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. η τρομοκρατία αποτελεί μια πολύ ε, βασική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Δηλαδή στην Αίγυπτο έχουμε ε, τρομοκρατικές ε, δράσεις όχι μόνο από την ίδια την μουσουλμανική αδερφότητα αλλά και από άλλες οργανώσεις που συνεργάζονται με τη μουσουλμανική αδερφότητα που απειλούν τον Αιγυπτιακό λαό και μέσα στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια και σε όλες τις περιφερειακές σε όλε τι περιφέρειε τη χώρα αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα, στο επίπεδο δηλαδή της βίας. Έτσι λοιπόν ε, το κράτο ε, τη Αιγύπτου έχει ξεκινήσει μια ναι, ένα πόλεμο κατά της ε, τρομοκρατίας δεν είναι η μόνη χώρα που βιώνει ένα τέτοιο μεγάλο κύμα τρομοκρατίας υπάρχουν πολλές άλλες χώρες ε, στην ε, Μέση Ανατολή και βέβαια μιλάμε και για την Αφγανική Ήπειρο που εδώ υπάρχουν πολλές οργανώσεις οι οποίες έχουν προβεί όχι μόνο σε τρομοκρατικές πράξεις αλλά και σε κλίματα πολέμου, σε εθνοκάθαρση και άλλες, άλλα τέτοια ε, αδικήματα. Δηλαδή δεν μιλάμε εδώ μόνο για την Αίγυπτο, μιλάμε για το σύνολο μιας, ε, ε, μιας περιοχής, δηλαδή χώρες, μια σειρά από χώρες τόσο της νοτίου Μεσογείου αλλά και της βορείου Μεσογείου που απειλούνται από τέτοιες ε, τρομοκρατικές ε, πράξεις ε, και γνωρίζουμε βέβαια τέτοιους είδους οργανώσεις δεν θέλουν την επιβολή ενός κράτους δικαίου και της δημοκρατίας αντιθέτως καταπολεμούν την ίδια την επιβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση αλλά νομίζω πως υπάρχει και μια ε, του ελπίδες. Ε, αυτή προέρχεται καταρχήν από το γεγονός ότι το νέο ή το Σύνταγμα της Αιγύπτου το 2014 έχει θέσει ε, ιδιαίτερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι το πρώτο Σύνταγμα το οποίο ποινικοποιεί τα βασανιστήρια, το οποίο θεσπίζει την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και προβλέπει και την θρησκευτική ελευθερία, ενώ προβλέπει ότι τον επιβάλλεται η κατάσταση συναγερμού στη χώρα ε, για περισσότερο από τρει μήνε μόνο με τη συνένεση του Κοινοβουλίου. Και, αυτό, και γι' αυτό δεν έχει επιβληθεί αυτή τη στιγμή. Ε, γιατί ακριβώ χρειάζεται κοινοβουλευτική συνένεση. Επίση, εάν ε, συγκρίνουμε τα δύο συντάγματα, αυτό εδώ δηλαδή το 2014 και εκείνο της μουσουμαλική αδερφότητας το 2012, θα δούμε μεγάλε διαφορέ. και για παράδειγμα, σε όλο το Σύνταγμα του 2012 δεν αναφέρονται εδώ μία φορά η, λέξη ανθρώπινα δικαιώματα και μάλιστα καταργούσε την ισότητα μεταξύ των ανδρών και των γυναικών ε, και ήταν υπέρ για παράδειγμα το Σύνταγμα ε, της δυνατότητας να υπάρχει ε, γάμος ακόμα και για παιδιά ε, νέα χρονών, με κορίτσια νέα χρονών. Με το νέο λοιπόν ε, Σύνταγμα έχουμε μια πολύ, μα πραγματικά πολύ βελτιωμένη εκδοχή που σέβεται τις βασικές αρχές, τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και ε, κάτι επίσης το οποίο είναι ελπιδοφόρον για το μέλλον είναι το γεγονός ότι η ε, Αιγυπτιακή κυβέρνηση ε, αποφάσισε και δεσμεύτηκε να εφαρμόσει την, τις συστάσεις του Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατά την τελευταία γενική κατά την τελευταία περιοδική αναθεώρηση και έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει 438 ε, τέτοιε συστάσει από σύνολο των 3.000. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τη μετώπιση των ε, βασανιστήριων, σε ό,τι αφορά ε, ε, την, το διοικητικό δίκαιο, το δίκαιο που διέπει τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και επίση. νομοθεσία, η, η ο τρόπος με τον οποίο υιοθετείται η νομοθεσία από την ε, Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Ε, καθώς υπάρχει ένα χρονικό όριο για την παρέμβασή μου, θα ήθελα να σας πω λοιπόν κλείνοντας ε, ε το τι συμβαίνει. Είναι, πρόκειται για έναν αγώνα ε, τον οποίο δίνουμε ε, ως ε, οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και όχι ένας αγώνας κατά της ε, κυβέρνησης αλλά ε, και ως προς το επίπεδο της κουλτούρας ε, των Αιγυπτίων. Δηλαδή, ε, πολλοί Αιγύπτιοι θεωρούν πως υπάρχει μια σχέση μεταξύ αυτής της ποινής και, του, και της Σαρία. Για παράδειγμα, ε, είχε ζητηθεί ε, κατά την ε, περίοδο ε, της κυβέρνησης του Μόρση να καταργηθεί η θανατική καταδίκη αλλά είχε αρνηθεί γιατί επρόκειτο θεωρούνταν ως Ισλαμικός νόμος. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει νέα δυνατότητα. Το ποινικό δικονομικό δίκαιο της Αιγύπτου τουλάχιστον προβλέπει τρία επίπεδα στο δικαστικό επίπεδο. Μετά δηλαδή από την πρώτη ε, καταδίκη έχουμε το ακυρωτικό δικαστήριο και μετά από το ε, ε, ακυρωτικό δικαστήριο περνάμε και πάλι στο ποινικό δικαστήριο. Δηλαδή υπάρχουν τρεις φάσεις αυτή η δικαστική διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει διάφορα χρόνια και υπάρχει πρόταση του κυρίου Σίση για αναστολή επιβολής της σχετικής ε, ποινής για 3, 5, 10 χρόνια προκειμένου να έχουμε κάποιο ε, ε, χρονικά περιθώριο τους ώστε να φτάσουμε στην κατάργηση του σχετικού άρθρου για την επιβολή της θαντικής ποινής και μέχρι τότε ενδεχομένως να υπάρξει και η σχετική ε, τελική απόφαση από την πλευρά του Μεγάλου Μουφτή. Ε, αγωνιζόμαστε κατά ανθρώπινα δικαιώματα, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και νομίζω πως ε, η Αίγυπτος θα καταφέρει στο μέλλον να δημιουργήσει ένα πραγματικό κράτος δικαίου που θα σέβεται ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Χαφέζα Μπουσεντά. Τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Μπαχέλντιν Χασάν. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε εδώ για μία ανταλλαγή απόψεων για το τι συμβαίνει στην Αίγυπτο ε, σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε έναν κοινό ε, φίλο με τον αδελφό μου, ο οποίος είναι ο ιδρυτής του κίνηματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ε, Αίγυπτο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι το Σύνταγμα εγγυάται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Άρα έκρινε ότι πρέπει να συνταχθεί ένας νόμος που να προστατεύει τους Αιγύπτιους πολίτες κατά των βασανιστήριων. Τι συνέβη σε αυτόν την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή ανακρίνεται και εκείνος και οι δύο δικαστές που συνέδραμαν σε αυτό το εγχείρημα και ε, η εταιρεία του, το δικηγορικό γραφείο του που, είναι, ε, που λειτουργεί εδώ και 74 χρόνια θεωρείται παράνομο δεν είναι ύποπτος τρομοκράτης, τον ξέρετε, πολλοί από εσά δεν είναι καν Ισλαμιστής, είναι κοσμικός. Και τώρα ε, τίθεται το ερώτημα τι συμβαίνει στην ε, Αίγυπτο πολεμάμε κατά όλων των κοσμικών. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Πολυτεχνείο, στο Πανεπιστήμιο του Πολυτεχνείου, η Ένωση των Φοιτητών παρετήθηκε μετά την ε, δολοφονία του Ισλάμ Ατίτο, ενός συμφοιτητή από τις ε, ε, δυνάμεις ασφαλείας. Το Υπουργείο Εσωτερικών είχε πει τότε ότι ήταν ε, υπέτειος για τη δολοφονία του συνταγματάρχη Βαέλ Ταχούν τον Απρίλιο του 2015 και έκτοτε, είχε, ε, και έκτοτε κρυβόταν στην έρημο έξω από το Κάιρο. Όμως ε, αυτόπτες μάρτυρες τον είδαν στο κάμπους του Πανεπιστημίου όπου συμμετείχε στην εξεταστική περίοδο. Εκεί μπήκαν δύο άνθρωποι που πήραν ε, την ταυτότητά του και τον συνόδευσαν εκτός ε, του Πανεπιστημίου. Έκτοτε οι μάρτυρες καθώς και, τη, και οι υπεύθυνοι της φοιτητική Ένωσης δεν είχαν νέα του και έχει εξαφανιστεί. Μετά το Υπουργείο Εσωτερικών την επόμενη μέρα ανακοίνωσε το θάνατό του. Αυτό μας δείχνει τι έχει γίνει η Αίγυπτος. Έχει γίνει μια δημοκρατία του τρόμου και λείπει εκλείπει ε, απόλυτα ένα καθεστώς ελέγχων και ισορροπιών. Το δικαστικό σύστημα έχει πολιτικοποιηθεί και ελέγχεται από δυνάμεις ασφαλείας. Και θεωρώ ότι δεν υπάρχουν ε, δεν υπάρχουν ε, εγγυήσεις, συνταγματικές ε, ε, εγγυήσεις έχουν παγώσει και υποσκάπτονται και από την εκτελεστική και από την δικαστική εξουσία. Επιπλέον, οι βουλευτικές εκλογές έχουν αναβληθεί πάρα πολλές φορές. Συνεντίε. Ο βασιλιάς ο Απτουλάχο δεύτερος της Ιορδανίας ε, πρόσφατα στο CNN είπε ότι το Συριακό καθεστώς ε, χτυπούσε οποιονδήποτε άλλο εκτός από την Άισις. Κατά τον ε, βασιλιά Απτουλάχ, η Συριακή κυβέρνηση χρειαζόταν μια τέτοια δύναμη. Μια δύναμη εκεί η οποία να είναι ακόμα χειρότερη. Όμως ο βασιλιάς της Ιορδανίας δεν αναφέρθηκε στην, στις ομοιότητες με άλλες αραβικές κυβερνήσεις όπως αυτή της Αιγύπτου η οποία βάλει κατά των αντιφρονούντων οποιοδήποτε προσανατολισμού. εκμεταλλεύονται τις τρομοκρατικές ενέργειες για να εξασφαλίσουν την αποδοχή και σιωπή της διεθνούς κοινότητας. Και έχουν επιβάλει δρακόντια ε, νομοθετικά μέτρα για να καταπολεμήσουν οποιοδήποτε αντιφρονούντα είτε είναι κοσμικός είτε Ισλαμιστής. Αυτές η αυτή η υπερβολική τακτική έχει δημιουργήσει ένα πολιτικό περιβάλλον όπου επικρατεί η βία. Ένα κενό το οποίο συχνά καλύπτουν οι φωνές των εξτρεμιστών. Υπάρχει μία κλιμάκωση ακριβώς επειδή υπάρχει μεγάλη σιωπή, σιωπή των ε, ορθολογιστών οι οποίοι θέλουν να δράσουν με ειρηνικά μέσα, αλλά αντιμετωπίζουν τις συλλήψεις, την όχληση και τελικά τη δολοφονία. Η δολοφονία του, της ε, ακτιβίστριας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της Σεΐμα Αλ-Σαμπάχ, είναι ένα παράδειγμα της δολοφονίας των ε, μαρτύρων, των μεγάλων μαρτύρων και των ε, υπερμάχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εκατοντάδες άλλοι αντιμετώπισαν την ίδια τύχη. και πολλοί έχουν καταδικαστεί σε κάθυρξη. Πιστεύω ότι η ριζοσπαστικοποίηση θα οδηγήσει στο χάος πολύ συντομότερα από ό,τι περιμέναμε. Η ύπαρξη εξτρεμιστών και τρομοκρατών στην περιφέρεια χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση ως δικαιολογία για να προβάλλει αυτές τις ακραίες πολιτικές το δικαίωμα ελεύθερης και δίκαιης δίκης έχει καταπατηθεί και δυστυχώς έχουν επιβληθεί ποινές κάθυρξης πολλών ετών ή ε, ισοβίων. Το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών μιλά για δίκες οι οποίες είναι παροδία δίκης. Έχουν επιβληθεί ποινές κάθυρξης κατά πολλών κοσμικών και Ισλαμιστών ακτιβιστών και πολλές ε, ε, φορές κρατούνται για παράλογα μεγάλα χρονικά διαστήματα. Παράλληλα, ε, υπάρχει έλλειψη αμεροληψίας και οι δικαιοδοτικές αρχές δεν είναι ανεξάρτητες, κάτι το οποίο δείχνει την αποτυχία τους. Το κράτος δικαίου στην, ε, στην Αίγυπτο είναι κάτι το ολοένα και πιο απόμακρο. Τον Απρίλιο του 2015 το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο ενέκρινε την ποινικοποίηση των ε, απεργιών και επέβαλε κυρώσεις κατά των απεργούντων των δημοσίων υπαλλήλων επιβάλλοντάς τους να συνταξιοδοτηθούν. Αυτή είναι η ερμηνεία του δικαστηρίου της ε, Σαρία. Από τον Ιούλιο του 2013 υπήρξε μία βελτίωση ως προς τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για τις γυναίκες και των δικαιωμάτων, και τα, των, δικαιωμάτων των κοπτών, αλλά τίποτα ε, δεν έχει βελτιωθεί. Ε, το δικαίωμα και η ελευθερία του συνέρχεστε έχει καταπατηθεί, καθώς και τα δικαιώματα των μη κυβερνητικών, καθότι στοχοποιούνται και τους επιβάλλονται έρευνες, απαγορεύεται να ταξιδέψουν μέλη των ΜΚΟ και υποβάλλονται σε συκοφαντική δυσφήμιση. Και αυτό εκεί όπου ζουν, εκεί όπου εργάζονται και φυσικά δεν έχουν δικαίωμα να ταξιδέψουν. Από τον Ιούλιο του 2013 πολλοί υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταδικαστεί σε πολιετή κάθυρξη, ενώ ένας ε, ακτιβιστής σκοτώθηκε, κάτι το οποίο είναι κάτι το ε, παράλογο μετά από το άνοιγμα των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την έναρξη των ε, κινημάτων υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο 30 χρόνια πριν. Το κοινό φοβάται και δεν μπορεί να εκδηλωθεί. Επικρατεί απόλυτη σιωπή. Από τον Ιούλιο του 2013 όλοι όλοι οι νέοι ηγέτες, κοσμικοί βέβαια, της ε, Επανάστασης του 2011, έχουν καταδικαστεί σε πολιετή κάθυρξη και σε πολλούς έχει επιβληθεί και ισόβια κάθυρξη. Μιλώ για ε, νέους ακτιβιστές, δεν μιλώ καν για Ισλαμιστές. Πολλοί αρθρογράφοι έπρεπε να επιλέξουν είτε να μείνουν στη χώρα τους είτε να φύγουν από αυτήν καθώς και πολλοί καλλιτέχνες και υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φαίνεται ότι δρούν υπόγεια και έτσι μπορούν μέρα με τη μέρα να επιδράσουν στη δράση των φιλελεύθερων ακτιβιστών η Αίγυπτος κινείται πολύ μακριά από τον, τη διαδικασία εκδημοκρατισμού. Έχουν αναβληθεί κατ' επανάληψη βουλευτικές εκλογές και δημιουργείται ένα κλίμα τρόμου Δυστυχώς ε, δεν διενεργούνται ε, εκλογές και όσοι θέλουν να υποβάλουν υποψηφιότητα αποθαρρύνονται για κάτι τέτοιο. Και από ό,τι φαίνεται, ακόμα και οι εκλογές στα συνδικάτα έχουν ε, απαγορευτεί. Δυστυχώς ούτε η εκτελεστική εξουσία ούτε η δικαστική δεν ε, υπόκειται στη λογοδοσία. Δεν έχουμε καμία επιλογή επιτάπητος. Και δεν τηρούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα. No Δεν υπάρχουν επιλογές. Η μόνη επιλογή ήταν πριν και μετά την Αραβική Άνοιξη. Τώρα όμως μιλάμε για βραχυπρόθεσμη σταθερότητα ή παγκόσμια σταθερότητα. Δεν θα υπάρξει καμία νίκη στην καταπολέμηση της σε αυτή την περιοχή, αν δεν δούμε τις ρίζες της κακοδαιμονίας. Εάν δεν λάβουμε υπόψη τα ακραία θρησκευτικά κινήματα και τους ε, κυβερνητικούς θεσμούς. Από τον Ιανουάριο του 2011 η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές είπε ότι δεν θα αποστρέψει το βλέμμα της όσον αφορά τις ε, μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι θα εμείνει στις ευρωπαϊκές αξίες. Αναρωτιέμαι κατά πόσο οι αρχές και αξίες αυτές διέπουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πολλών εθνικών κοινοβουλίων σε σχέση με τις παραβιάσεις αυτές, αλλά οι δηλώσεις αυτές δεν έχουν καμία επίπτωση στην ε, πραγματικότητα, στις καθημερινές ε, δράσεις, ε, στην καθημερινή δράση στην Αίγυπτο. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ροντρίγκε είναι η πρώτη που έχει ζητήσει το λόγο από τους συναδέρφους. Κάποιος άλλος, ο κύριος και επίσης. Ναι, και εσείς. Εντάξει, κυρία Ροντρίγκης όμως πρώτα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω πορτογαλικά, αν μου επιτρέπετε. Ευχαριστώ για τους ε, συναδέλφους, ε, ευχαριστώ τους συναδέλφους και ευχαριστώ και τους παρεμβαίνοντες που μας ε, μίλησαν για το τι συμβαίνει στην Αίγυπτο επειδή είμαι αντιπρόεδρος της Euromed για θέματα πολιτισμού. Έχω παρακολουθήσει την κατάσταση αυτή. Έχω τρεις βασικές ανησυχίες και στους τέσσερις. Μιλήσατε γι' αυτό, μιλήσατε για τη θανατική ποινή την ελεύθερη κυκλοφορία και την ε, παρέμβαση των ΜΚΟ, καθώς και το δικαίωμα στον πολιτικό ακτιβισμό. Πρόκειται για ένα δικαίωμα και εγώ ήμουνα ακτιβίστρια όταν ήμουν νέα. Δεν μπορώ να φανταστώ μια χώρα χωρίς πολιτικό ακτιβισμό, ιδιαίτερα στα πανεπιστήμια. Ένας τομέας που με απασχολεί είναι η βία κατά των γυναικών. Υπάρχει η αρχή της μη διάκρισης και της ε, ισότητας δικαιωμάτων. Αυτό το εξασφαλίζει το Σύνταγμα, αλλά βλέπουμε ότι έμπρακτα δεν ισχύει, δεν εφαρμόζεται. Θα ήθελα να σας ακούσουμε περισσότερο για τα γενικά αυτά δικαιώματα, κατά πόσο δηλαδή υπάρχει εγγύηση αυτών των δικαιωμάτων υπέρ των γυναικών. Εγώ προσωπικά πιστεύω και ίσως θα μπορούσατε να με διαφωτίσετε. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει ποινικοποίηση της φυσικής βίας κατά των γυναικών. Το άρθρο 268 και το 306 όπως έχουν διαμορφωθεί θα πρέπει να μας οδηγήσουν στην καταπολέμηση ιδιαίτερα της οικογενειακής βίας και να εξευρεθούν στρατηγικές. Υπάρχουν. Θα προσπαθήσω να μην ε, επεκταθώ γιατί έχω πολλές ερωτήσεις. Πώς ε, μπορεί ο σύζυγος να επιβάλλει αυτού του είδους την πειθαρχία στη σύζυγό του και επίσης τι γίνεται ως προς τα εγκλήματα τιμής είναι ένα θέμα που μας απασχολεί μέσα στα πλαίσια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πώς η συζυγική βία δεν αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον ποιδικό κώδικα, τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση. Πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε τα δικαιώματα των γυναικών να τύχουν σεβασμού και ως προς τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο συμμετείχαν στην εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Ε, <clears throat> Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Οι πληροφορίες αυτές που μας έδωσαν οι δύο προσκεκλημένοι μας εννοείται ότι δεν μας οδηγούν σε υπερβολική αισιοδοξία. Ακούσαμε ότι οι θεσμικές εγγύησεις προβλέπονται, αλλά ο δεύτερος προσκεκλημένος μας είπε ότι έχουν παγώσει. Οπότε το Αιγυπτιακό κράτος από τη μια έχει δημιουργήσει το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από την άλλη μεριά όμως δεν λειτουργεί. Οπότε, ρωτάω, εσείς που γνωρίζετε καλά την πραγματικότητα στην χώρα, αυτή η διαδικασία πώς θα μπορούσε να συνεχιστεί, τι πιθανότητες υπάρχουν να βγει η χώρα από αυτού του είδους το διέξοδο. υπάρχουν συνταγματικές αρχές από τη μια, αλλά από την άλλη η πραγματικότητα δείχνει κάτι εντελώ διαφορετικό. Πιστεύω λοιπόν ότι η απόσυρση ας πούμε της ε, αποστολής παρατήρησης των εκλογών είναι κάτι συμβολικό. Θα έλεγα ότι είναι δύσκολο να δεχτούμε μια διαδικασία η οποία λαμβάνει χώρα κάτω από τέτοια κατάσταση όπου οι διεθνείς ε, οργανισμοί δεν το δέχονται. Έπειτα αυτοί οι ακτιβιστές της πλατείας Ταχύρ μεταξύ αυτών υπήρχε και μία γυναίκα η οποία βραβεύτηκε με το βραβείο Ζαχάροφ από εμάς. Και αυτή βρίσκεται μεταξύ αυτών που καταδικάστηκαν. Και τρίτον, τρίτο ερώτημα, υπάρχει ένα τεράστιο ανθρωπιστικό πρόβλημα που έχει να κάνει με την μετανάστευση μετά ακριβώς την Αραβική Άνοιξη. Όχι ας, σαν συνέπεια, αλλά επειδή στη Λιβύη ιδιαίτερα δεν λειτουργούν οι κρατικοί θεσμοί. Αλλά και η Αίγυπτος είναι χώρος από τον οποίο περνούν όλοι αυτοί οι μετανάστες. Μετανάστες που έρχονται από την Ερυθρέα, τη Σομαλία και που είναι και αυτοί θύματα της μετανάστευσης. Το Αιγυπτιακό κράτος λοιπόν κάνει κάτι για να αποφύγει αυτή την κατάσταση. Στα μέσα ενημέρωσης συχνά μας παρουσιάζουμε πολύ τραγική κατάσταση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Δεμασμάκερ. Ευχαριστώ πολύ. Ολλανδικά θα μιλήσω. Πρώτα απ' όλα θέλω κι εγώ να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας για την ενημέρωσή τους. Η Αίγυπτος είναι μια σημαντική χώρα στην περιοχή, έχει σημαντικό ρόλο να παίξει για την ασφάλεια πρώτα απ' όλα. Η καταπολέμηση του φονταματαλισμού λοιπόν, της ριζασπαστικοποίησης σε ολόκληρη την περιοχή κατά του φανατισμού του θρησκευτικού είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και η Αίγυπτος λοιπόν απειλείται από την τρομοκρατία και είναι και θύμα της τρομοκρατίας. Οπότε λοιπόν βρίσκω ελπιδοφόρο το ότι η κοινωνία των πολιτών στην Αίγυπτο με αλληλεγγύη αντέδρασε στον θάνατο 21 κοπτών τον Φεβρουάριο στη Λιβύη. Είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα αυτό. Βέβαια, το καθεστώς θέλει να αποφύγει την απειλή της τρομοκρατίας. Δεν μπορεί όμως αυτό να αποτελεί άλοθη ώστε να παραβιάζει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα συστηματικά. Ανησυχούμε λοιπόν όλος ιδιαίτερος, μετά από αυτό που ακούσαμε και σήμερα, όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο. Μας ανησυχεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται ελευθερίες. Μετά την πτώση του Μουμπάρακ, του Μόρση, πώς πιέζονται οι ελευθερίες αυτές. Ζητάμε λοιπόν, κάνουμε έκκληση στην κυβέρνηση της χώρας να προστατεύσει τις ελευθερίες και να τηρήσει όσον αναφέρονται στο Σύνταγμα για τις ελευθερίες. Τα λόγια είναι καλά, αλλά τα λόγια αυτά πρέπει να γίνονται και πράξεις. Δεν έχει νόημα να έχουμε ένα πολύ όμορφο σύνταγμα αν δεν τίθεται σε εφαρμογή. Η πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει λίγα αποτελέσματα από ό,τι φαίνεται. Οπότε το ερώτημα είναι εμείς πώς μπορούμε να επηρεάσουμε περισσότερο την κατάσταση. Θα ήθελα λοιπόν μία απάντηση ε, να πάρω στην ερώτηση αυτή. Και πρέπει και να αναρωτηθούμε επίσης πώς εμείς συγκεκριμένα μπορούμε να βοηθήσουμε. Σκέφτομαι για παράδειγμα το πρόβλημα που παραμένει για την υπερβολική βία από πλευρά τη αστυνομία. Στις διαδηλώσεις έχουμε πάντα νεκρούς. Στις φυλακέ. επίσης υπάρχει κακομεταχείριση που καταλήγει σε θανάτους μερικέ φορές. Πώς λοιπόν μπορεί να ελεγχθεί αυτή η κατάσταση. Με κατάρτιση των αστυνομικών. Πώς λοιπόν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει περισσότερο ώστε να υπάρξει κάποια αλλαγή νοοτροπίας. Έπειτα, η ελευθερία του τύπου και η ελευθερία έκφρασης είναι κάτι που με απασχολεί και εμένα πολύ. Ήμουν δημοσιογράφος, δεν θεωρώ ότι είμαι κανένας κακοποιός. Η δημοσιογραφία δεν είναι έγκλημα. είδαμε ότι έγιναν συλλήψεις δημοσιογράφων. Ο Πέτερ Γκρέστερ της Αλτζαζίρα ελευθερώθηκε, ένα χρόνο όμως πέρασε στη φυλακή. Φοβούμε λοιπόν ότι η ελευθερία αυτή τελικά μείωσε το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας απέναντι στις παραβιάσεις της ελευθερίας του τύπου στη χώρα. Τι λέτε εσείς για αυτήν την πίεση από πλευράς ε, της διεθνούς κοινότητας. Και τελειώνω με αυτό που είπα στην αρχή. Η διεθνής κοινότητα στηρίζει σιωπηρά την κυβέρνηση της σημερινή της Αιγύπτου επειδή πρόκειται για έναν σταθερό εταίρο στην περιοχή. Από φόβο δηλαδή, μήπως δημιουργήσει αλλιώς αποστεθαροποίηση στην περιοχή. Ποια είναι η γνώμη σας από αυτού. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Εκ μέρους των Πρασίνων, ο κύριος Μπίχνερ. Ευχαριστώ πολύ. Μου δίνετε το λόγο και ευχαριστώ πολύ για τη διοργάνωση αυτής της ε, αυτή τη συζήτηση την οποία θεωρώ πραγματικά απαραίτητη. Ε, το ερώτημά μου αφορά ειδικότερα ε, στη σχέση μεταξύ την, ε, της κανονικών δικαστηρίων και στρατιωτικών δικαστηρίων. Και θα αναφερθώ ειδικότερα εδώ στις έξι εκτελέσεις που έλαβαν χώρα στις 17 Μαΐου. Από ό,τι κατάλαβα λοιπόν ε, ε, προηγουμένως είχαν ε, εξαφανιστεί τα εν λόγω αυτά πρόσωπα χωρίς να γνωρίζει κανείς πού βρίσκονται, σε ποια φυλακή κρατούνται. Άρα λοιπόν ε, πρόκειται για μια διαδικασία η οποία ε, έλαβε χώρα εκτός των κανονικών δικαστικών διαδικασιών της χώρας. Ε, πρόκειται δηλαδή για την εξαφάνιση αυτών των προσώπων, δηλαδή ε, μιλάμε ότι δεν γνώριζε κανείς που βρίσκονται. Τα δικαστήρια που τους δίκασαν ήταν στρατιωτικά δικαστήρια, οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω, τέτοιου είδους ψευδονομικές διαδικασίες λαμβάνουν συχνά χώρα στη, ε, στην Αίγυπτο. Ε, και ένα ακόμα ερώτημα, τέτοιου είδους έξοδικαστικές αν θέλετε εκτελέσεις καταδικασμένων. Ε, είναι συχνό φαινόμενο. Ε, λαμβάνουν χώρα μόνο σε στρατιωτικό πλαίσιο. Τι συμβαίνει. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, θα δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, στην κυρία Νίκολα Κιλχό. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και ευχαριστώ πολύ τους προσκεκλημένους από την Αίγυπτο που μας ενημέρωσαν για την τρέχουσα κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο. Σύμφωνα με τα όσα μας είπατε, εξακολουθεί να είναι ανησυχητική. Όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα λοιπόν, η κατάσταση είναι ενισχυτική και εμείς παρακολουθούμε από κοντά όχι μόνο εδώ, από εδώ που βρισκόμαστε με τέτοιες ανταλλαγές απόψεων όπως η σημερινή, αλλά συναντιόμαστε και με συναδέρφους σας στην υπηρεσία μας, αλλά και επιτόπου η αντιπροσωπεία μας παρακολουθεί στενά την κατάσταση και συνομιλεί με την κοινωνία των πολιτών και την αντιπολίτευση. Προσπαθούμε λοιπόν έτσι να έχουμε μια πλήρη εικόνα και από την κυβέρνηση εννοείται, αλλά και από άλλους παράγοντες στην Αίγυπτο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, οι ομιλητές μας να αντιδράσουν, παρακαλώ, να απαντήσουν. Ε. Σύντομα, δύο-τρία λεπτά, παρακαλώ. Δύο-τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Θα ε, αρχίσω με τον κύριο Χασάν καλύτερα. Ε? Παρακαλώ. Μια που εκείνος μίλησε δεύτερος, θα μιλήσει τώρα πρώτος. Δύο-τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων. Προσπαθώ, θα προσπαθήσω να σχολιάσω δύο-δυόμιση λεπτά Βέβαια είναι mission impossible. Δεν είμαι πολύ σύντομο. Τηλεγραφικά θα σας απαντήσω. Διάφορες ερωτήσεις ετέθησαν μεταξύ άλλων και για τα δικαιώματα των γυναικών. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Υπάρχει πολιτική βούληση για μια όμορφη παρουσία και εγώ είμαι πολύ περήφανος για τα όσα αναφέρονται γραπτά αλλά βλέπω ότι τελικά οι Αιγύπτιοι πολίτες έχουν τέτοια δικαιώματα όχι μόνο για να τα δείξουν σε εσά όταν πηγαίνετε εκεί ως ε, αποστολές. Αυτό που βλέπετε εσείς δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Ακόμα και οι νέοι νόμοι και οι τροπολογίες που περνάνε καθημερινά παραβιάζουν το ίδιο το πνεύμα του κεφαλαίου αυτού του συντάγματός μας που αναφέρεται στα δικαιώματα των γυναικών. Χτες μόλις ο πρόεδρος ενός από τα φιλελεύθερα κόμματα έκανε μια δήλωση και ζήτησε από τον πρόεδρο να διαγράψει το κεφάλαιο το σχετικό κι όμως τέτοια γίνονται. ζήτησε να διαγραφεί να διαγράψει το ίδιο το κοινοβούλιο, γιατί είμαστε από αναβολή σε αναβολή, οπότε βλέπετε ότι τελικά οι ίδιοι νόμοι οι οποίοι προτείνονται παραβιάζονται στη συνέχεια. Οπότε τι νόημα έχει. Αυτό είναι ένα από τα κύρια προβλήματα λοιπόν που έχουμε στην Αιγυπτιακή πολιτική σήμερα. Κάτι άλλο που ρωτήσατε είχε να κάνει με τις εξοδικαστικές δολοφονίες. Δεν πρόκειται μόνο για τον Άχδα και τον Ράμπτα. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις και ο που ήταν ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν πήγε να κάνει τίποτα άλλο, λουλούδια πήγε να αφήσει. Ένα άλλο θέμα είναι πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τη ποιοντατού είναι η ηθική της, φωνή, φωνή της ηθικής όπως είπα και νωρίτερα, υπογραμμίζει όλο και περισσότερο το θέμα του σεβασμού των ευρωπαϊκών αξιών. Συνεπώς, πιστεύω ότι υπάρχει κοινό συμφέρον μεταξύ της Αιγύπτου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τέρη. Η Αίγυπτος πρέπει να πετύχει στον αγώνα της υπέρ της σταθερότητας κατά της τρομοκρατίας, αλλά στην πραγματικότητα δεν επικεντρώνεται τόσο σε αυτά. Ο πραγματικός αγώνας πάει οπουδήποτε αλλού, εκτός από αυτά. Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε ότι όλοι οι μη θρησκευτικοί ηγέτες έχουν φυλακιστεί από τρία χρόνια μέχρι ισοβίως. Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε ότι όπως Αλμαμπατστά δολοφονούνται, πώς βοηθάει αυτό τη σταθερότητα της Αιγύπτου, την ευημερία των Αιγυπτίων, πώς βοηθάει τη σταθερότητα της περιοχής στη Λιβύη, στο Ιράκ και αλλού. Φοβάμαι ότι αυτά είναι γεγονότα. Συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο όπως το Ιράκ και η Λιβύη, αν συνεχίσει η Αίγυπτος έτσι. Δεν βοηθάει τη σταθερότητα της χώρας. Αν το πιστεύει αυτός κάποιο, κάποιος αυτό είναι ψευδέστηση. Αυτό είναι που προσπαθήσαν και ο Ασάντ και οι υπόλοιποι στις άλλες χώρες με τα αποτελέσματα που ξέρουμε. Ξέρουμε τι θα γίνει αν συνεχίσουμε έτσι. Αν συστηματικά κάνουμε άλλα πράγματα, προσωποποιούμε τους θεσμούς. Και κυρίως αυτή την περιοχή που είναι γεμάτη εξτρεμιστές, ξέρουμε που θα οδηγήσει. Έτσι θα διαδοθεί περισσότερο η τρομοκρατία και όχι το αντίθετο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει ο επόμενος προσκεκλημένος μας. Ευχαριστώ για όλα τα ερωτήματα που θέσατε. Ε, πραγματικά ήταν σημαντικά και μας δίνουν την ελπίδα ότι υπάρχει μια διεθνής ε, κοινότητα η οποία γνωρίζει ε, το τι συμβαίνει στην Αίγυπτο και είναι σε θέση να βοηθήσει τους, ε, τον λαό της Αιγύπτου σε ό,τι αφορά τον, το κράτος δικαίου. Ναι, υπάρχουν ε, μία σειρά από περιπτώσεις που αφορούν την κοινωνία των πολιτών και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουμε σε μία λύση. Για παράδειγμα, στην περίπτωση ε, εκείνου του δημοσιογράφου όπου αναφέρθηκε ότι δεν ήταν η σφαίρα που τον σκότωσε, δεν προχώταν από αστυνομία, αλλά τελικά εμείς επιμείναμε ότι πράγματι ήταν από αστυνομία και ζητήσαμε, αξιώσαμε να υπάρξει μια σωστή έρευνα και τελικά τι έγινε, η αστυνομία έδωσε στο Γενικό Εισαγγελέα ε, το όνομα του αστυνόμου, ο οποίος σκότωσε τον λογοπρόσωπο και βρίσκεται τώρα σε φάση δίκης. Ναι, υπάρχουν κάποιες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά σε όλο τον κόσμο υπάρχει ακριβώς ένας αγώνας για την τήρησή τους. Αλλά εγώ διαφωνώ ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση στην Αίγυπτο και αυτό γιατί ο λαός της Αιγύπτου θέλει, πραγματικά επιθυμεί, να γίνει κάτι τέτοιο και δεν φοβούνται αφού έχουν λάβει χώρα δύο επαναστάσεις. Και θα ήθελα να απαντήσω σε δύο ε, πιο συγκεκριμένα ζητήματα. Πρώτα, σε ό,τι αφορά βία εις βάρος των γυναικών. Αυτή την περίοδο ε, ε συνεργαζόμαστε ως κοινωνία των πολιτών σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης ε, για αυτό το ζήτημα. Δηλαδή πρέπει μετά από την ε, συνταγματική αναθεώρηση, έχει υπάρξει λίγος χρόνος για να ε, ε, προβούμε στι αντίστοιχε τροποποιήσει στο ποινικό μας δίκαιο και ούτω καθεξής. Δηλαδή δεν είμαστε πραγματικά στην ίδια διαδικασία όπως ήταν τότε με τον Χουσέιν, τώρα με τον Μπασάλα Σάντε. Δεν, δεν βρισκόμαστε στην ίδια φάση. Έχουμε ένα σύνταγμα στην Αίγυπτο και είμαστε ω ιδιακό λαό σε θέση να το το, το, να το εφαρμόσουμε στην πράξη, όχι να μείνει δηλαδή επί χάρτου μόνο το Σύνταγμα. Και χρειαζόμαστε κάποιο χρόνο για να τροποποιήσουμε την, ε, την νομοθεσία μας. Και, ε, και στο πλαίσιο των ε, ε, βουλευτικών εκλογών, ε, στι οποίε ήμουν και εγώ υποψήφιο, ναι, ακούσαμε το τι έγινε. Ότι δηλαδή ο τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η, η εκλογική διαδικασία ε, ε, δεν ακολούθησε τα όσα ε, προέβλεπε και το Σύνταγμα. Ε, εν πάση σε ό,τι αφορά τις εργασίες που κάνουμε σε ό,τι αφορά τους μετανάστες. Ναι, πρόκειται για μια επικίνδυνη κατάσταση για όλες τις χώρες. Υπάρχουν δηλαδή κάποια πρόσωπα τα οποία και από το χώρο της τρομοκρατίας τα οποία έρχονται στη Μεσόγειο. Και πραγματικά όποιος νομίζει ότι δεν υπάρχει ε, τομοκρατία προφανώς δεν υπάρχει ένας, ε, μια, ένας αγώνας τον οποίο την αστυνομία και ο στρατός και θα σας δώσω κάποια ε, στοιχεία 700 ε, αστυνομικοί έχουν σκοτωθεί ε, σε περίοδο τριών μηνών. Μιλάμε για οπλοπολιβόλα τα οποία φέρνουν οι ε, τρομοκράτες μαζί τους ε, περνώντας μέσω για παράδειγμα των ε, συνόρων με το Σουδάν, με τη Λιβύη έρχονται και από αλλού και ε, πρόκειται πραγματικά για έναν, έναν αγώνα, έναν πόλεμο τον οποίο έχουμε στη χώρα μας κατά της τρομοκρατίας και προσπαθούμε και με αυτήν την μεταρρύθμιση του συντάγματος να σεβαστούμε και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι, ο πρόεδρος έχει ένα όρομα ότι δηλαδή θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα ε, στους κοινωνικούς και οικονομικούς ε, στόχους αλλά από την άλλη πλευρά προσπαθούμε να του τονίσουμε ότι το ένα πολύ σημαντικό είναι βέβαια και η σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ένα τελευταίο σημείο. Ποιο είναι ο ρόλο που μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια στρατηγική σχέση μεταξύ Ένωση και Αιγύπτου και υπάρχουν πολλοί τρόποι με το οποίο μπορεί να μα βοηθήσει. Τεχνική υποστήριξη για τους, ε, τι νομικέ αρχέ, ε, το ε, γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα και ούτω καθεξής. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική υποστήριξη η οποία ε, γίνεται μέσω του, της εταιρικής ε, σχέσης ε, και κατά τα τελευταία 14 χρόνια. Επίσης θα πρέπει να είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε τις μη κυβερνητικέ οργανώσει και στο πλαίσιο τη νομοθεσία που διέπει τι μη κυβερνητικέ οργανώσει, προκειμένου αυτό ο νέος νόμος να επιτρέπει να υπάρχουν και να είναι πιο φιλελεύθερο ε, τηρώντας πρώτα το, το, το Σύνταγμα και το κράτος δικαίου. Ε, αυτή είναι η ελπίδα μας να υπάρξουν αυτές οι εξελίξεις στο μέλλον και ελπίζουμε ότι και εμείς θα μας ε, υποστηρίξετε ώστε να επιτύχουμε να είμαστε μια χώρα που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Ως ήθιστε στην Επιτροπή μας θα δώσουμε το λόγο και στον πρέσβη της Αιγύπτου. Είναι ο κύριος Αντέλ Ιμπραχήμ, ο οποίος είναι αναπληρωτής επικεφαλής αποστολών. Έχει το λόγο. Τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πράγματι σύντομος. Η Αίγυπτος, τα γαλλικά, έτσι. Δεν θα μιλήσω αραβικά. Τα τελευταία χρόνια όντως υπήρχαν δυσκολίες, αλλά πάλι καλά τα καταφέραμε τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Αποφύγαμε τα χειρότερα, διατηρώντας αυτά που θεωρούμε σημαντικά και ο λαός και η κυβέρνηση, που είναι ο δρόμος προς τη δημοκρατία. Αξιότιμοι ευρωβουλευτές, εκτιμούμε όλους ιδιαίτερως το ενδιαφέρον που δείχνεται για, την εξέλιξη, για τις εξελίξεις στη χώρα μας. Όπως επίσης και το ενδιαφέρον που έχει δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα για την ε, Αίγυπτο. Όμως πρέπει να σας ε, μεταφέρω την αίσθηση που επικρατεί στον Αιγυπτιακό λαό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει την κυβέρνηση πολύ περισσότερο από ό,τι τη συνοδεύει προς τη δημοκρατία. Πρόεδρε, παρακολούθησα τη συνεδρίαση της υποεπιτροπής σας πριν από δύο χρόνια εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επενθυμίζω ότι τότε είχαν επικρίνει οι ευρωβουλευτές και είχαν εκφράσει την ανησυχία τους για την πολιτική την εποχή εκείνη των αδερφών μουσουλμάνων. Η κατάσταση ήταν σοβαρή, όπως είπανε, και χαρακτηριζόταν από συγκρούσεις στους δρόμους της Αιγύπτου και προετοίμαζαν το δρόμο για αμφίλιο πόλεμο κάτι το οποίο συνέβη αργότερα σε πολλές χώρες στην περιοχή. Πρόεδρε, θέλω να υπογραμμίσω εδώ το πόσο λεπτό είναι το ζήτημα, πόσο λεπτή είναι η κατάσταση σήμερα στην Αίγυπτο. Αστυνομικοί δολοφονούνται κάθε μέρα, ο στρατός ε, αγωνίζεται κατά της τρομοκρατίας στο Σιναή. Προσπαθούμε να τηρήσουμε τι αρχέ τις οποίε πιστεύει η Αίγυπτος. Η καταπολέμηση τη τρομοκρατία δεν πρέπει να γίνεται σε βάρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμω πρέπει να υπάρχει μια δυσκολία, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο σήμερα. Μια δημοκρατία δεν φτιάχνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Υπάρχει μια μετάβαση προ τη δημοκρατία, η οποία δεν ήταν τόσο εύκολη ούτε τόσο γρήγορη στις χώρες Ανατολικής Ευρώπης μετά τον ψυχροπόλεμο. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Και όσον αφορά τη θανατική ποινή, έχουμε την πεποίθηση ότι η συζήτηση για το κατά πόσο πρέπει ή δεν πρέπει να υπάρχει είναι περίπλοκη και μακρά. Παρ' όλα αυτά, η Αιγυπτιακή κυβέρνηση ή κυβερνήσεις της Αιγύπτου πάντα ήταν ανοιχτές κάθε φορά που συζητιόταν το θέμα αυτό, για τη θανατική ποινή δηλαδή στα διεθνή φόρα. Λαμβάνουμε υπόψη μας ότι παραμένει μία ποινή που στηρίζεται από ένα μεγάλο μέρος του Αιγυπτιακού λαού. Πρόεδρε, η θανατική ποινή αποτελεί μέρος του ποινικού κώδικα της Αιγύπτου. Όσο ισχύει αυτό, κάποια εγκλήματα θα τιμωρούνται με τη θανατική αυτή ποινή. Τέλος, θέλω να σας διαβεβαιώσω για το ότι τα λάθη των αστυνομικών δυνάμεων έχουν αναγνωριστεί από την κυβέρνηση και δεκάδες αστυνομικοί έχουν βρεθεί πρώτη δικαιοσύνη. Με ποινέ βαριέ. Τέλος, Πρόεδρε, για τη δικαστική εξουσία. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειε, αλλά δεν δέχομαι να μιλάτε για μεροληψία της δικαιοσύνης. Ευχαριστώ πολύ. Merci. Ε. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ για την παρέμβασή σας, κύριε Πρέσβη. Για τη θανατική ποινή θέλω να αναφέρω ότι η Νεμπράσκα κατάργησε χτες τη θανατική ποινή. Κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μας είναι ένα πάρα πολύ θετικό νέο. Όπως το είπα και στην αρχή, αυτή είναι η άποψή μας για Όλοι σε αυτό θέλετε να αντιδράσετε για την Εμπράσκα. Για, για πείτε μας. Θέλω να πω ότι αν μια συζήτηση στην κοινωνία των πολιτών καταλήγει στην κατάργηση και συμβεί και αυτό και στη χώρα μου σε 30-40 χρόνια, θα το δεχτώ. Εγώ προσωπικά είμαι κατά τη θανατική ποινή. αλλά όσο ο νόμος λέει ότι υπάρχει, ισχύει. Είμαι εγώ προσωπικά. Από το 81, από τότε που καταργήθηκε στη Γαλλία. Ευχαριστούμε πολύ για την αντίδρασή σα αυτή λέει ο πρόεδρο. Η συζήτηση αυτή ήταν πολύ πλούσια. Ακούσαμε διαφορετικές απόψεις και τους συναδέρφους και τους προσκεκλημένους και όλους. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα και για την ποιότητα των παρεμβάσεών σας. Πριν ολοκληρώσουμε, θέλω να σας πω ότι η επόμενη συνεδρίαση της υποπιτροπής μας θα λάβει χώρα στις 16 και 17 Ιουνίου 2015 βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε.